και είναι η δήλωση της Κομισιόν για την κρίση σε γεωργικούς τομείς εκτός του γαλακτοκομικού τομέα. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Φίσερ Μπέλ που είναι μαζί μας και σας δίνω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, καταρχάς σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να έρθω εδώ και να εξηγήσω την ε, σημερινή οικονομική κατάσταση στον γεωργικό τομέα. Τα οικονομικά, η οικονομική κρίση και η χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε φυσικά και τη γεωργία. Ε, είχαμε ύφεση και μείωση της ζήτησης, εξέλιξη των ε, συναλλαγματικών ισοτιμιών, δύσκολη πρόσβαση σε πιστώσεις και όλα αυτά είχαν προφανώς μια επίπτωση στις γεωργικές τιμές και στο εισόδημα των γεωργών. Οι επίσημε εκτιμήσει για το γεωργικό εισόδημα θα είναι στη διάθεσή μα στο τέλος τη εβδομάδας. Αλλά περιμένουμε ότι το εισόδημα θα μειωθεί ουσιαστικά μέσα στο 2009 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά το 2008 δεδομένης της εξέλιξης ε, στο κόστος παραγωγής ε, και, των, και δεδομένων των αλλαγών στις γεωργικές τιμές. Μετά την αρχική μείωση που παρατηρήσαμε το 2008, αυτή η νέα μείωση των γεωργικών τιμών και των εισοδημάτων των γεωργών θα εξουδετερώσει κάποιες αυξήσεις που προήλθαν που αφορούσαν κάποια γεωργικά προϊόντα και που ξεκίνησαν να παρατηρούνται από το καλοκαίρι του 2007. Θα ήθελα να μιλήσω για διάφορους τομείς. Καταρχάς για τα Δημητριακά, Πρόεδρε. Το 2008 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των τιμών των σιτηρών. Ίσως λόγω καλής οδειάς. Παρόλα αυτά, οι τιμές τους ε, τελευταίους ε, μήνες αυξήθηκαν, ιδίω για το σιτάρι και το καλαμπόκι. Λόγω αυτών των εξελίξεων δεν θα ήταν σωστό σε αυτή τη στιγμή να λάβουμε εξαιρετικά μέτρα όπως ε, το άνοιγμα της ε, ε, παρέμβασης για το καλαμπόκι, ούτε να δώσουμε εξαγωγικές επιστροφές. Η κατάσταση είναι κατά τη διαφορετική για το κρυθάρι με μειωμένες εξαγωγές και χαμηλές εσωτερικές τιμές. Αλλά η παρέμβαση, όπως ξέρετε, έχει αρχίσει, έχει ανοίξει και αυτό θα πρέπει να βοηθήσει τις αγορές. Στον τομέα του χείριου κρέατος η κατάσταση είναι εύθραυστη. Η οικονομική κρίση έπληξε σε μια χρονική στιγμή όπου δεν είχαμε ανακτήσει πλήρη πλήρως από τις ε, προβληματικές ε, στιγμές του 2007. Οι τιμέ ε, φέτος είναι χαμηλότερε από το 2008 και παράλληλα ε, ας δείξουμε και λίγη αισιοδοξία. Οι ελεύθερε τιμές είναι πιο σταθερές από ότι το 2007 και 2008. Και παρότι οι εξαγωγέ ήταν χαμηλές και χαμηλότερες από τα επίπεδα του 2008, θα είναι μεγαλύτερες Παρ' όλα αυτά, το, τις εξαγωγές του 2007. Συνολικά, λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος για να βάλουμε περαιτέρω μέτρα αγορέα σε αυτή τη φάση. Θα παρακολουθήσουμε όμως την κατάσταση εκ του σύνεγγης. Τα προκυπευτικά τώρα. Η οικονομική κρίση οδήγησε σε χαμηλότερη εσωτερική κατανάλωση και επίσης υπάρχουν και κάποιες μειώσεις ε, σε κάποιες αγορές λόγω εξαγωγών. Αυτό επηρέασε τις τιμές ε, των παραγωγών για τα οποροκυπευτικά. Δεδομένων όμως των χαρακτηριστικών του τομέα, αποφασίσαμε στην τελευταία μεταρρύθμιση των οποροκυπευτικών να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ε, του τομέα και πώς το αποφασίσαμε, τι αποφασίσαμε να κάνουμε, να καταστήσουμε πιο ελκυστικές τις οργανώσεις των παραγωγών και να τις καταστήσουμε υπεύθυνε για τη διαχείριση των κρίσεων. Οι οργανώσεις των παραγωγών σήμερα αποτελούν το 40% του συνολικού, της συνολικής παραγωγής ε, φρούτων και λαχανικών και μπορούν να ανταπεξέλθουν γιατί είναι πιο δυνατές οικονομικά. Φυσικά η σημερινή κρίση δεν αναγνωρίζει εθνικά σύνορα. Το 2007, ε, στη μεταρρύθμιση που κάναμε, προβλέψαμε ε, ότι θα υπάρχουν κάποια κίνητρα για τις οργανώσεις των παραγωγών για να αντισταθούν. Επίσης, τους δώσαμε νέα εργαλεία διαχείρισης της κρίσης. Παραδείγματος χάρη τη δυνατότητα να μην υπάρξει εσοδιά που συνοδεύει τις παραδοσιακές αποσύρσεις. Επίσης υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που επιτρέπει τους παραγωγού αυτού παραγωγούς αυτούς να επηρεάσουν την αγορά και να τη σταθεροποιήσουν. Όμως πρέπει να υπάρχει δράση από κάτω προς τα πάνω. Η Κομισιόν όμως δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ενθαρρύνω τις οργανώσεις παραγωγών και μάλιστα ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να δημιουργήσουν περισσότερες οργανώσεις. Θα πρέπει να δούμε τους αριθμούς ε, που έχουμε στα διάφορα κράτη-μέλη, τους αριθμούς οργανώσεων παραγωγών. Αν ανταγωνίζονται οι οργανώσεις ε, μεταξύ τους δεν έχει νόημα, αντί να ανταγωνίζονται το λιανεμπόριο. Ελαιόλαδο. Οι τιμές αυτές έφτασαν, ε, χτύψαν ρεκόρ πριν από τέσσερα χρόνια λόγω των κλιματικών συνθήκων. Και μετά από τρεις ε, ικανοποιητικές οδιές, η οικονομική κρίση τελικά βαθμία οδήγησε στην πτώση των τιμών και τελικά σε πολύ χαμηλές τιμές. Γι' αυτό η Κομισιόν ε, επανεργοποίησε φέτος την ιδιωτική αποθεματοποίηση και είδαμε ότι η αγορά αντέδρασε πάρα αυτά. Και τελικά οι τιμές ανέκαμψαν και σταθεροποιήθηκαν. Παρά λοιπόν τις καλές προβλέψεις για τη σοδιά, τέταρτη καλή σοδιά, η, τα αποθέματα στην αρχή της σοδιάς ήταν χαμηλά. Και θεωρούμε ότι τελικά θα ανακάμψει και η κατανάλωση. Συνολικά λοιπόν υπάρχουν κάποια δειλά δείγματα ανάκαμψης. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση και να δράσουμε όταν απαιτείται. Είναι μια γρήγορη επισκόπηση αυτή κάποιων βραχυπρόθεσμων θεμάτων. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι έχουμε και βραχυ... μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη θεώρηση. Παραδείγματο χάρη την κατανομή της προστιθέμενης αξίας στην διατροφική αλυσίδα, αντιμετώπιση της αστάθειας των τιμών κτλ. Όλα αυτά τα σημαντικά θέματα θα τα ξαναδούμε, Πρόεδρε. Τώρα το λόγο Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Εκ μέρου των πολιτικών ομάδων για την κοινοβουλευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο κύριος Ντες για δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Στα προηγούμενα χρόνια αλλά και φέτος οι γεωργοί διαμαρτυρήθηκαν και στις Βρυξέλλες κιόλας. Όχι όμως μόνο η γαλακτοπαραγωγή, είναι γεγονός ότι και άλλες και άλλοι κλάδοι έχουν πληγεί από την κρίση εκτός από τους γαλακτοπαραγωγούς, οι χειροτρόφοι, οι εκτροφείς πουλερικών, αλλά και ορισμένοι που σπέρνουν και καλλιεργούν δημητριακά, έχουν ζήσει και καλύτερες χρονιές. Και γι' αυτό τώρα διαμαρτύρονται. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι καλό που σήμερα ρίχνουμε φως στην κατάσταση και αυτών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Όπως είπατε κύριε Επίτροπε, η οικονομική, χρηματοπιστωτική κρίση έφτασε πλέον και σε ολόκληρη τη Γεωργία και την έπληξε. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουμε. Συζητώντας επί τόπου με πληγέντες γεωργούς, ακούω συχνά να μου λένε ότι τα καταφέρνουμε να βαδίζουμε στις αγορές, εκτός βέβαια από καταστάσεις όπου διαγράφονται πολύ δύσκολες όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια για προϊόντα αλλά και φέτος για το γάλα. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι γεωργοί και οι αγρότε γενικά είναι η συνεχή γραφειοκρατική επιβάρυνση από πλευρά ευρωπαικη Ένωση. Εμεί λένε θέλουμε να βγαίνουμε έξω στα χωράφια μα και στα λιβάδια μα, να φροντίζουμε τα ζώα μα. όχι να καθόμαστε όλη την ημέρα να συμπληρώνουμε έντυπα και βιβλία. Για ολόκληρους αιώνε μπόρεσαν οι αγρότες μας να παράγουν τρόφιμα, να γίνονται οι δημοπρατήσεις, να αυξάνεται η παραγωγικότητα των ζώων. Σήμερα τους παραφορτώνουμε με γραφειοκρατία. Βλέπω τώρα ότι οι Υπουργοί Γεωργίας εγκύπτουν <clears throat> στην μελέτη του θέματος σε μια προσπάθεια να μειώσουν την γραφειοκρατία. Ας κάνουν ό,τι μπορούν, γιατί αυτό που θέλουμε οι αγρότες μας είναι να παράγουν τρόφιμα καθαρά, υγιεινά για μισό δισεκατομμύριο εν τέλει συμπολίτε μα. Ε, ε, και Δημοκράτες, ο κύριος Ντεκάστρο για δυόμιση λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ακόμα μια φορά συζητούμε την κρίση στο γεωργικό τομέα. Τους τελευταίους μήνες το Κοινοβούλιο εκφράστηκε πολλές φορές ε, πάνω στις δυσκολίες ε, που έπληξαν πάρα πολύ ειδικά τον τομέα του γάλακτος και ζητήσαμε από το, την Κομισιόν και το Συμβούλιο να παρέμβουν κατεπηγόντως. Είχαμε αποτελέσματα παρότι ήταν μερικά, αλλά με βάση τέτοιες πρωτοβουλίες ε, τελικά δημιουργήθηκε ένα ταμείο 300 εκατομμύρων ευρώ για να αντιμετωπίσουμε την επίγουσα κατάσταση. Η κρίση λοιπόν ε, που καταρχάς έπληξε το γάλα τώρα ε, απλώνεται γρήγορα και σε άλλους τομείς. Ε, ανισχυτικά σημάδια βλέπουμε στο σκληρό σύτο, στο ελαιόλαδο, στα οπροκυπευτικά, όπως είπε και η Επίτροπος Φισερμπόλ. Όπως και για το γάλα, αντιμετωπίζουμε πίζουμε ένα διαρθρωτικό φαινόμενο που συνοδεύει τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω της μείωσης της ζήτησης και της καθίζησης των αγορών. Η κρίση λοιπόν δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα όπως δείχνουν και τεράστιες διαμαρτυρίες που ε, υπάρχουν σε πολλέ περιφέρειες τη Ευρώπη. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι πραγματικά ανησυχητική και μα ανησυχεί το μέλλον συνολικά του τομέα, του γεωργικού τομέα. Γι' αυτό ακριβώ την τελευταία συνεδρίαση, την 1η Δεκεμβρίου τη Επιτροπή Γεωργία, ομόφωνα αποφασίσαμε να καλέσουμε εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε τι γίνεται με την κρίση τη γεωργία. Ε, και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα, την κρίση που αντιμετωπίζουν οι επιμέρους τομείς της γεωργίας. Καταρχάς, η Κομισιόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέτρα που έχει στη διάθεσή της για να σταθεροποιήσει την αγορά και να ε, τονώσει την ζήτηση και την κατανάλωση. Επίσης, όμως, θα πρέπει να στραφούμε προς το μέλλον. Να δώσουμε διασφαλίσει ότι η κοινή γεωργική πολιτική θα εξακολουθήσει να είναι μια σημαντική ευρωπαϊκή πολιτική και που θα ε, αφορά τα συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων πολιτών και όλων ε, ε, των, ε, περιφερειών. Από το βορρά στο νότο, από το, τις ε, βαλτικές περιοχές ως την Κύπρο. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να επιταχύνουμε τις ε, δράσεις μας και για να ε, δείξουμε ότι διδαχθήκαμε από τα μαθήματα του παρελθόντος. Δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Θα πρέπει να διορθώσουμε μια κατάσταση η οποία μπορεί πραγματικά να εξοκύλει. Θα θέλαμε να μα δοθούν απαντήσει. Και ενδεχομένω, αν υπάρχει κάτι καινούργιο να μα πει η Κομισιόν, είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Δεκαστρο, ήσασταν και ακριβεί στον χρόνο. Τώρα για την ομάδα των φιλελευθέρων, η κυρία Χάρκιν για ένα λεπτό παρακαλώ. Thank you, Madam President. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο για την κατάσταση που μας περιέγραψε. Θέλω να εστιάσω την προσοχή μου σε ένα τομέα που μπορούμε πράγματι να δράσουμε. Αυτό έχει να κάνει με το χαμηλό επίπεδο απαγορευμένων γενετικά τροποποιημένων ε, προϊόντων σε ζωοτροφές που επηρεάζει ιδιαίτερα την αγορά. Έθεσα ένα ερώτημα προς τον κύριο Μπαρόσο και είπε ότι η Κομισιόν ενέκρινε τρία προϊόντα γενετικά τροποποιημένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές αλλά ακόμα δεν έχουμε προλάβει χώρες όπως η Βραζιλία η οποία έχει επιταχύνει τα συστήματα έγκρισης και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εύκολα αυτό το πρόβλημα. Ξέρουμε ότι είναι χαμηλό το επίπεδο κερδοφορία στις αγροτικές αγορές και αυτό το οποίο περιμένουν όλοι οι γεωργοί είναι να μειωθεί το κόστος των εισρωών επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δράσει ταχαίω για να εξασφαλίσει την ε, ε, έγκριση ε, προϊόντων ζωοτροφών. Όταν δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα, αυτό μας θέτει σε μειονεκτική θέση. 23 εκατομμύρια χαθήκαν για αυτόν τον λόγο στην Ιρλανδία. Το επίπεδο της χαμηλής παρουσίας γενικά τροποποιημένων προϊόντων θα υπάρχει πάντα. Χρειάζεται μια ταχεία διαδικασία έγκρισης για αυτό χρειαζόμαστε τις τεχνικές λύσεις. Ξεπεράστε το χρόνο σα όμως και δεν πρέπει να γίνει το ίδιο με του επόμενου συναδέλφου. Ε, τώρα εκ μέρου τη ομάδα των Πρασίνων, ο κύριο Χάουσλινγκ για δύο λεπτά παρακαλώ. Κυρία Επίτροπε, κυρίε και κύριοι, η απάντηση που δώσατε ήταν σύντομη. Δεν άκουσα να προσφέρετε ιδέες για λύσεις. Όντως έχουμε κρίση στο γάλα, έχουμε κρίση στα δημητριακά. Έχουμε και συγκέντρωση στα οπροκυπευτικά και χάσαμε και 10% όλων των εκμεταλλεύσεων της χειροτροφίας τα τελευταία χρόνια. Αυτά δεν οφείλονται στην οικονομική κρίση, οφείλονται στο γεγονό ότι ο προσανατολισμό τη ε, αγροτική πολιτική τα τελευταία χρόνια ήταν εσφαλμένο. Μπορεί να πει κανεί ότι η φιλελευθερωποίηση απέτυχε, το άνοιγμα στην παγκόσμια αγορά δεν είναι λύση για την γεωργία. Θα πρέπει να αποφασίσουμε για τα επόμενα χρόνια προ τα πού θα κατευθυνθεί η γεωργία μα. Γι' αυτό χαιρόμαστε που δώσαν ένα ξεκάθαρο ε, σήμα οι υπουργοί στο Παρίσι για το που θα πάνε. Χρειαζόμαστε ασφάλεια σχεδιασμού και βιωσιμότητα. Και γι' αυτά εμείς επιμένουμε. Πέφτουν οι τιμές για τους γεωργούς, όχι όμως για τους καταναλωτές. Αυτό δείχνει ότι η γεωργική πολιτική εξυπηρετεί κυρίως τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρήσεων. Είπατε κι εσείς, κυρία Επίτροπε, σωστά, ότι πρέπει να ενισχύσουμε τον ρόλο των αγροτών. Αλλά εξακολουθείτε να μην δίνετε απάντηση στο πώς θα το κάνουμε αυτό. Αυτό σας ζητώ να πράξετε, να δώσετε απάντηση γιατί θα είναι κρίσιμο αυτό για τα επόμενα χρόνια. Οι αγρότες δεν μπορεί να υποβαθμιστούν μοναχά σε παραγωγούς βιολογικών καυσίμων. Πρέπει να έχουν ευρεία ποικιλία προϊόντων. Ασκείται πίεση στην υγειοργία. Αυτό θα οδηγήσει σε ελλείψεις ποιότητας, σε ακόμα περισσότερη εκβιομηχάνηση, άρα μικρότερη ποικιλότητα. Και μια εκβιομηχανισμένη γεωργία θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος με διοξίδια του άνθρακος και μεθάνιο. Από τη μια λοιπόν πληρώνουμε για να σώσουμε το κλίμα, από την άλλη μεριά κάνουμε την γεωργία μεγαλύτερο παραγωγό τέτοιων αερίων. Τα από τους συντηρητικούς ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι κατανοούμε τις ανησυχίες πολλών τομέων μέσα στη γεωργία και ίσως δίνουμε πολύ υπερβολική έμφαση για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του γαλακτοκομικού τομέα σε σχέση με του άλλου τομεί. Αυτοί όμω οι οποίοι ανεπλάξαν σε αυτή τη διαδικασία του γαλακτοκομικού τομέα ξέρουν δεν υπήρχε εναλλακτική λύση. Ευτυχώ έχουμε επιλύσει κάποια από τα καυτά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο τομέα αυτό και τώρα πρέπει να δώσουμε προσοχή και σε άλλου τομεί τη γεωργία. Αναφέραμε το θέμα των ε, ε, γεωργών που παράγουν σιτηρά που αντιμετώπισαν πάρα πολύ χαμηλές τιμές στην αγορά και η ε, παραγωγή πατάτας και μήλων στην περιοχή μου είχαν πάρα πολλά σημαντικά προβλήματα. Μπορώ να σας πω, να σας δώσω ένα μακρύ κατάλογο περιοχών όπου υπήρξαν προβλήματα. Αλλά θέλω να επανέλθω σε αυτό που είπε η κυρία Χάρκιν. Το κύριο πρόβλημα είναι η καθυστέρηση για να εγκριθούν ε, εισρωές για ζωοτροφές που βασίζονται σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία εισαγωγών ζωοτροφών για χείρους και για άλλα είδη για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Βρισκόμαστε σε ένα σοβαρό κίνδυνο αυτή τη στιγμή. Να πληγούμε από υπερβολική γραφειοκρατία και από νομοθεσία η οποία οδηγεί σε ασφυξία τους γεωργούς μας και ιδίω από την 1η Ιανουαρίου που θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα, το CPID, το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι απόλυτα άχρηστο και ανώφελο. Είμαστε έτοιμοι για αλλαγέ, αλλά αυτό που είναι απαραίτητο είναι να εξετάσουμε το αποτέλεσμα τη εφαρμογή τέτοιων αλλαγών στο παρελθόν. Γνωρίζω από την περιοχή μου ότι πολλοί κτηνοτρόφοι που εκτρέφουν πρόβατα και έγες φεύγουν πια από την κτηνοτροφία και τους τομείς αυτούς. Θα πρέπει να δούμε πώ υποστηρίζουμε του γεωργού και του κτηνοτρόφου. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο και να του διατηρήσουμε στη γη. Γιατί πολλοί από αυτού του τομεί είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι για το περιβάλλον και είναι η μόνη δραστηριότητα σε ορισμένε περιοχέ όπου δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατή δραστηριότητα. Πρέπει να του υποστηρίξουμε λοιπόν. Τώρα από την Ενωτική Αριστερά ο κύριος Λε Ιαρίκ για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, μας είπατε ότι η γεωργική κρίση είναι βαθιά. Αυτό το ξέραμε ήδη. Βεβαίω, οι μικροί γεωργοί και οι μεσαίοι γεωργοί πραγματικά δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Αλλά αυτό δεν είναι αποτέλεσμα τεχνικού προβλήματο. Είναι αποτέλεσμα τη δική σα πολιτική απελευθέρωση, την οποία τη ε, σπρώξατε ε, στα πλαίσια τη ΚΑΠΑ αρνείστε να υπάρχουν ελάχιστε τιμέ και είσαστε υπέρ των ελεύθερων συναλλαγών ε, και εναντίον της αρχή της προτίμηση. προτίμησης. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε εκ νέου ε, για την κοινή γεωργική πολιτική. Θα πρέπει να δούμε ότι η πολιτική αυτή έχει κάνει κοινοφελές έργο. Μία νέα ΚΑΠ θα πρέπει λοιπόν να είναι μια επισητιστική πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική και εδαφική πολιτική. Θα πρέπει να δούμε καταρχάς ποιοι είναι οι προσανατολισμοί. Ποια είναι ε, η κατεύθυνσή της πριν αποφασίσουμε για τα δημοσιονομικά ζητήματα. Ούτω ή άλλω, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αμείβονται με ελάχιστες εγγυημένε τιμές οι γεωργοί. Μία παραγωγική ε, γεωργία θα πρέπει να εξασφαλίζει απασχόληση, θα πρέπει να εξασφαλίζει την αρχή της επιστηστικής ασφάλειας ενάντια στους λοιμούς. Όλα δείχνουν σήμερα ότι η κοινωνική, περιβαλλοντική, η υγειονομική αποτελεσματικότητα βασίζεται σε μια γεωργία που στηρίζεται σε ανθρώπινες ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Μόνο έτσι νομίζω θα βγούμε από τη σημερινή γεωργία της κρίσης. Ο κύριος Φοντάνα για δύο λεπτά από την Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε. Η σημερινή κρίση που ζει ο κόσμος της Γεωργίας είναι το αποτέλεσμα της ε, γρήγορης επέκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια και κυρίως της πολύ γρήγορης παγκοσμιοποίησης των αγορών. Ο γεωργικός τομέας θα πρέπει να διαφυλαχθεί εφαρμόζοντας την αρχή της α, ίσης μεταχείρισης που δημιούργησε την Ευρωπαϊκή ε, Κοινότητα, άρθρο 31-38. Και ιδίως θα πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένους νομικούς κανόνες. Σε αυτόν τον τομέα, οι κανόνες που ε, ρυθμίζουν την παρέμβαση δεν μας δίνουν τις σωστές απαντήσεις δεν προστατεύουν τον Γεωργό. Σε μια στιγμή εξαιρετικά δύσκολη που εμπλέκει όλους τους τομείς τους γεωργικούς και κυρίως τα οποροκυπευτικά, παραδείγματο χάρη ε, μήλα ε, και ροδάκινα, ε, αντιμετωπίζετε πρόβλημα λοιπόν. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή μεταχείριση, κάτι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ή υπάρχει με πολύ περιορισμένο τρόπο. Είδαμε ότι η κρίση του γάλακτος και σήμερα ε, η κρίση των οβορκυπευτικών ε, επεκτείνεται. Σήμερα ε, νομίζω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να πάρει τις σωστές δράσεις, να υποστηρίξει τους γεωργούς και τις εκμεταλλεύσεις τους, οι οποίοι υποστηρίζουν την επικράτειά μας, κάτι που το ξεχνάμε συχνά. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά για να ουσιαστικά υποστηρίξουμε τις δικές μας παραγωγές και όχι τι ξένε παραγωγέ. Ιδίω στον τομέα των απορροκυπευτικών. Να έχουμε συγκεκριμένου κανόνε, του οποίου θα πρέπει να σέβεται ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε και να το επιβάλλουμε και στι τρίτε χώρε με τι οποίε έχουμε σημαντικέ ε, συναλλαγές, ούτως ώστε να έχουμε μία αγορά χωρί τρευλώσει. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω θα υποστηρίξουμε ουσιαστικά και την Ευρωπαϊκή Γεωργία και του Γεωργού. Ο για δύο λεπτά Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τομείς της αγροτικής οικονομίας δοκιμάζονται πραγματικά. Σιτηρά, ελαιόλαδο, φρούτα και λαχανικά, βαμβάκι. Θα ήθελα να σας πω κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αίσθημα οργής διακατέχει τους παραγωγούς ροδακίνων στην Ελλάδα, αρκεί να σας αναφέρω ότι 200.000 περίπου τόνοι κομπόστας είναι αδιάθετοι τη στιγμή που μιλάμε. Η κατάσταση στον τομέα των σιτηρών παραμένει απαιτεί κρίσιμη και απαιτεί να ενεργοποιηθεί άμεσα η δυνατότητα δημόσιας παρέμβασης στα κράτη μέλη. πρέπει να στηρίξουμε τα προϊόντα προστατευόμενης ε, ονομασίας προέλευσης καθώς και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης. κτηνοτροφία μεγάλη κρίση αναφερθήκαμε και ορθώς αναλάβαμε την πρωτοβουλία για την προστασία του, του γαλακτοκομικού τομέα. αλλά θέλω να σου πω ότι κτηνοτρόφοι στη βόρεια ελλάδα απέκτησαν το τελωνείο ε, των ευζώνων και ένα από τα μέτρα ένα από τα αιτήματα τα εύλογα αιτήματα τα οποία θέτουν είναι η αναγραφή της ονομασίας του τόπου προέλευσης στις συσκευασίες των γαλακτοκομικών προϊόντων. Και πράγματι, κατά τη γνώμη μου, η αναγραφή του τόπου προέλευσης προστατεύει και τους παραγωγούς αλλά και τους ε, καταναλωτές. Χρειαζόμαστε περαιτέρω μέτρα για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων τόσο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός, ε, σε τρίτες αγορές, εκτός Ευρώπης. Πρέπει να εξορθολογιστούν ακόμη περισσότερο οι αγορές, να παρακολουθήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο τη διαφάνεια της εφοδιαλιστικής αλυσίδας και να μειώθει οπωσδήποτε η ψαλίδα μεταξύ τιμών παραγωγού και τιμών καταναλωτή. Όπως είχα υποστηρίξει και στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2010, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρηθεί ένα ικανοποιητικό περιθώριο γεωργικών δαπανών στον προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών σε άλλους ε, γεωργικούς ε, τομείς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Παπαστάμκο. Τώρα συνεχίζουμε τους, ε, τις παρεμβάσεις. Ο κύριος Σταμπάτζη για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε όλη η ευρωπαϊκή γεωργία αντιμετωπίζει μια κρίση. Αυτό δεν αποτελεί τμήμα μονάχα της παγκόσμιας κρίσης και της μείωσης της έκτασης των αγορών στο εσωτερικό και το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι και απόρρια της μορφής που έλαβε η Ευρωπαϊκή Αγροτική πολιτική. Η νεοφιλελεύθερη αυτή πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει συμβάλει τα μάλα στην τωρινή κρίση. Αν τώρα ο αγροτικό τομέα έχει να αντιμετωπίσει τόσο σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά τα έσοδα των γεωργών, τι θα γίνει μετά από το 2013 όταν θα μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η υποστήριξη από τον αγροτικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο θεωρούν ότι είναι απαραίτητο. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η τροφοδοσία με τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω σε ό,τι αφορά το χείριο κρέα και το τομέα των οπροκυπευτικών. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι θέλετε να δώσετε περισσότερα χρήματα στι κοινέ οργανώσει αγορά αλλά αυτό δεν θα επαρκέσει για να επιληθούν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο αγροτικό τομέα. Επιπλέον, αν πάρουμε σαν παράδειγμα το βόλιο κρέα, η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι καθαρό εισαγωγέα. Επομένω, βρισκόμαστε στο έλεος τη διεθνού αγορά. Και έχει το λόγο για ένα λεπτό, παρακαλώ. ευχαριστώ. Εξετάστε τα μέτρα που λαμβάνει η ε, Βρετανική κυβέρνηση για το κατόφλι εισοδήματος. Ένα τέταρτο όλων των ε, Βρετανών γεωργών πέφτουν στην κατηγορία αυτή. Και θα έπρεπε να ασχολούμαστε εδώ όχι μόνο για μια αγροτική προσέγγιση, αλλά μια συνολική προσέγγιση. Γιατί οι καταναλωτές αυτό, αυτό που θέλουν είναι τρόφιμα καθαρά, υγιή, τα οποία να παράγονται κοντά στον τόπο που μένουν. Η επισήμανση των τροφίμων με ετικέτες για να γνωρίζουν από πού προέρχεται είναι σημαντική. Έχουμε ήδη κανόνες που επιβάλλουν την ετικετοθεσία σε προϊόντα σχετικά με την χώρα προέλευσή τους. Γιατί να μην επεκταθεί και να περιληφθούν και τα βασικά συστατικά μεταπημένων τροφίμων. Ας, ε, ε, ας αλάβουμε τις απαραίτητες αποφάσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εδώ και πολλά χρόνια μετά από διαδοχικές αλλαγές της κοινή αγροτικής πολιτικής βλέπουμε συνέχεια τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί και εμείς καταθέτουμε εναλλακτικές προτάσεις. Κανείς δεν θέλει να μας ακούσει βέβαια και σήμερα αντιμετωπίζουμε και πάλι μια κατάσταση ολέθρια η οποία λαμβάνει η χώρα στην Πορτογαλική Γεωργία. Θέλουμε να σας προειδοποιήσουμε για τις συνέπειες της φιλελευθερωποίησης του Διεθνού εμπορίου των αγροτοτροφημικών προϊόντων. Η γεωργία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν να είναι απλώς μια βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα. Θα πρέπει να μείνει έξω των διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για να μην είναι θύμα των ε, κερδοσκοπικών ενεργειών σε επίπεδο χρηματιστηρίων ή σε επίπεδο αγορών. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ε, τροφιμική ασφάλεια και να δώσουμε αξιοπρέπεια σε αυτούς οι οποίοι δουλεύουν την υγιή και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε σωστά θέματα όπως αυτό το γαλακτοκομικό ποσοστό. Υπάρχουν εξάλλου ιδιαίτερε συνθήκες στις χώρες της Νότιας Ευρώπης που θα πρέπει να τύχουν σεβασμού γιατί είναι οι χώρες οι οποίες παράγουν προϊόντα μεγάλης ποιότητας όπως είναι ε, τα προκυπευτικά το κρασί, το λάδι, αλλά και προϊόντα ε, ζωικά τα οποία είναι μεγάλη σημασία για άλλες χώρες. Επειδή λοιπόν είναι υψηλό το κόστος των εισρώων στη γεωργία, του φυσικού αερίου, πετρελαίου, του ηλεκτρισμού κτλ. θα πρέπει να έχουμε πολιτικές οι οποίες θα υποστηρίξουν τους γεωργούς με πολιτικές οι οποίες θα διασφαλίσουν την απασχόληση στον αγροτικό χώρο δίνοντας έμφαση στην οικογενειακή γεωργία και δίνοντας τη δυνατότητα να μπορέσουν να ορθοποδήσουν οι περιφερειακές και τοπικές παραγωγές. Οι γεωργοί πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι παράγουν τα απαραίτητα για την υγεία μας και τη διατροφή μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έγνιου έχει το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ. Well, President, looks as I've... Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, Νομίζω ότι είμαι ένας από τους οπαδούς της κυρίας Χάρκιν, γιατί τονίζω τα προβλήματα που έχει η αγορά ζωοτροφών μπορεί να υπάρξουν ίση, ίσως ίχνο, ίχνη μη γενετικών γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Και αν βρεθούν τέτοια ίχνη δεν μπορεί να εκφορτώσει κανείς τις ζωοτροφές. Μπορεί να σημαίνει ότι έχουμε απώλεια λοιπόν τελωνιακών εσόδων. Αλλά έχουμε και μεγάλη διαταραχή της αγοράς όταν τα φορτηγά γυρίζουν άφορτα και χωρίς αποτέλεσμα στις ε, στη, στο, στο χώρο προέλευσής της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, θεωρήσει ότι η παρέμβαση γενικά τροποποιημένων οργανισμών στο, στον Αβόστο μπορεί να είναι αποδεκτή. Αλλά συγχρόνως στις ΗΠΑ εγκρίνονται νέες ποικιλίε γενετικά τροποποιημένου αραβόστου που όλο και περισσότερο θα εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λαμβάνει υπόψη ότι μπορούν μέσα στα μεγάλα φορτία αραβοσίτου να υπάρξει ανάμειξη γενικά τροποποιημένων οργανισμών που οδηγεί σε απόρριψη, σε μη έγκριση αυτών των φορτίων. Αλλά υπάρχουν και πριονίδια, υπάρχουν νεκρά έντομα, υπάρχουν ε, ε, μεταλλικά αντικείμενα μέσα στα φορτία που δεν μπορούν να αποφευχθούν πολλές φορές. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να απορρίπτεται η είσοδο των φορτίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει μεγάλα προβλήματα και για τους παραγωγούς και για τους καταναλωτές αυτών των προϊόντων. Αυτή είναι μια κατάσταση που οδηγεί σε υψηλή σε υψηλέ τιμέ στον τομέα τη ξενοτροφία. Η Κομισιόν θα πρέπει να αντιμετωπίσει με ένα πιο λογικό και πρακτικό τρόπο με το να έχει ένα μεγαλύτερο επίπεδο ανοχή για τι ε, προσμίξει γενετικά τροποποιημένων ουσιών. Λαβία για δύο λεπτά επίση, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επίτροπο για την ανάλυση που μας έκανε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι σε ορισμένους παραγωγικούς τομείς ενσκύπτει σήμερα μια κρίση που θέτει ένα αμφιβόλο την ε, βιωσιμότητα της γεωργίας σε ορισμένες περιοχές της μεγάλης μας Ευρώπης. Ιδίως η κρίση η οποία πλήττει τους τελευταίους μήνες το σκληρό σύτο. Ε, οδήγησε τις τιμές του σκληρού σύτου σε τιμές ανεπαρκείς για να καλύψουν τα κόστη, το κόστος παραγωγής και σε ορισμένε ε, περιοχές της Ευρώπης μειώνονται οι σπαρμένες ε, επιφάνειες. Ε, ιδίως σε περιθωριακές ε, περιοχές που δεν υπάρχουν εναλλακτικέ καλλιέργειε. Επίσης η επίτροπο μίλησε για το προκυπευτικά. Μίλησε για τη νέα ΚΟΑ. Αφήνει τους, τις οργανώσεις των παραγωγών να διαχειριστούν την κρίση. Φυσικά, οι πόροι που τους δίνονται στα, στο εσωτερικό των ε, επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι περιορισμένοι, που σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν για να παρέμβουμε σε περίπτωση διαρθρωτικής κρίσης ε, και τόσο εκτεταμένης όπως αυτή που ζούμε σήμερα. Μπορούν ενδεχομένως να καλύψουν τα τρέχοντα έξοδα, όπως, όπως για την ε, όπως για αυτές τις περιπτώσεις που είπατε, όταν υπάρχουν μικρο ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Ε, σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν ε, τις επιπτώσεις μια τόσο ευρείας κρίση όπως αυτή που ζούμε. Το ίδιο ισχύει και για το ελαιόλαδο και για άλλα προϊόντα. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση είναι σημαντικό να τονίσουμε και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πακέτο από προτάσεις και να διατυπώσει μία διαρθρωμένη πρόταση που θα αφορά όλους τους τομείς που ε, που σε καμία περίπτωση δεν, ε, δεν είδαν ε, μέτρα στοχευμένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αντίθεση με αυτό που συνέβη στο Γάλα. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο αγροτικός τομέας δεν είναι στις δυσκολίες της γενικής οικονομίας. Αλλά είχαμε την ευκαιρία ήδη στο παρελθόν να τονίσουμε τα προβλήματα που έχουν οι γαλακτοπαραγωγοί. Τότε πολλοί από εμά Τονίσαμε ιδιαίτερα το γεγονό ότι η κρίση αυτή είχε επεκταθεί και σε άλλου γεωργικού τομεί. Η κατάσταση λοιπόν η οποία ισχύει για το σύνολο τη γεωργία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχουν χαμηλέ τιμέ που είναι η πηγή του προβλήματο και πολλέ αγροτικέ εκμεταλλεύσει βρίσκονται πια κάτω από το όριο της ε, αποδοτικότητας και της κερδοφορίας. Αυτό, αυτό είναι και αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο κατανέμεται η προσθέμενη αξία στον αγροτικό τομέα. Πρέπει να υπάρχει μια επανεξισορρόπηση μέσα στην νομοθεσία για να υπάρχει και μεγαλύτερη δυνατότητα διαπραγμάτευση των γεωργών έναντι των αγοραστών. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η υπόσκαψη τη αντιγωνιστικότητα των γεωργών που δεν μπορούν να καλύψουν το, το χάσμα που του χωρίζει από άλλου παραγωγού σε άλλα τμήματα του κόσμου. Επομένως, δεν μπορεί να βασίζεται μια απάντηση μονάχα στα κρατημέρια, πρέπει να υπάρχει συνολική αντιμετώπιση. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι το σημείο αυτό είναι σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Είναι μια ευκαιρία να κατανοήσουμε όλοι ότι υπάρχει ένας ε, κίνδυνος και μια κρίση όχι μόνο στο γαλακτοκομικό τομέα αλλά σε όλη τη γεωργία. Αυτό είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό για όλους τους γεωργού να μπορέσουμε να συζητήσουμε για την κατάστασή τους και να προχωρήσουμε σε κάποια εξέβριση λύσεων. Η χρηματοοικονομική κρίση έχει χτυπήσει ιδιαίτερα του γεωργού, Είναι από τους ε, πιο πληγέντε και η κατάστασή του είναι πράγματι ζωφερή η κρίση αυτή και τα δημόσια ελλείμματα έχουν σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν ελλείμματα σε επίπεδο νοικοκυριών. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε μια καταστροφή αν δεν κάνουμε τίποτα και υπάρχουν πραγματικά προβλήματα σε ανθρώπινο επίπεδο. Μέσα από αυτή την κρίση όμως υπάρχει και μια δυνατότητα να βελτιώσουμε τα πράγματα και αυτή η ευκαιρία πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Για να γίνει κάτι τέτοιο η Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσει την διαταραχή της ισορροπίας στον τομέα αυτό και δεύτερον θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για τους γεωργούς το οποίο επιτρέπει να υπάρχει μια αυτορύθμιση από τη μεριά των ίδιων των γεωργών τρίτον οι νομικές αρμοδιότητες των συνεταιρισμών γεωργών πρέπει να βελτιωθούν επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε τη χρήση ανανεώσιμων ενεργειών από τους γεωργούς μέσα σε μια ρύθμιση <clears throat> της αγοράς για να βελτιώσουμε τα προβλήματα αυτά. Πέμπτον, δεν θα πρέπει να υπάρξει μονάχα κατάλυση της γραφειοκρατίας, αλλά μία απλοποίηση όλων των διαδικασιών. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτή την κρίση η οποία, και τις ευκαιρίες που υποκρύπτονται σε αυτή την κρίση για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους γεωργούς μας να μην είναι αυτοί τα θύματα της ε, οικονομικής κρίσης αλλά να μπορέσουν μέσα από τον κατάλογο μέτρων της ε, Επιτροπής που θα συζητήσουμε στην Αρμόδια Επιτροπή να βελτιώσουν τη θέση τους. λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Θέλω να σας χαιρετήσω για την παρουσία σας και πάλι στην Ολομέλεια που είναι μια σταθερή παρουσία σας σε όλη την ε, διάρκεια αυτής της θητείας παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε μεταβατική φάση η Επιτροπή. Βέβαια η Γεωργία δεν μπορεί να περιμένει τα καπρίσια της πολιτικής. Οι Γεωργοί περιμένουν από εμάς να τους δώσουμε μια λύση για τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Ξέρουμε ότι η οικονομική κρίση έφυξε επίσης σε μεγάλο βαθμό και τη Γεωργία. Όχι μόνο στον τομέα της γαλακτοκομικής παραγωγής όπως τα μέσα ενημέρωση μπορεί να δίνει την εντύπωση ότι ισχύει, αλλά και σε άλλους τομείς γεωργίες. Στα οποροκυπευτικά, στο ελαιόλαδο, στα σιτηρά. Όλα αυτά επλήγησαν ιδιαίτερα και όχι μόνο το γάλα το τελευταίο καιρό και αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια αύξηση των συντελεστών κόστους στην παραγωγή βοήου κρέατος. Για τα προκυπευτικά φαίνεται ότι η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη τη στιγμή που υπάρχει ένα άνοιγμα της αγοράς για τα προϊόντα του Μαρόκου μέσα στη νέα συμφωνία η οποία, της οποίας επίκειται η έγκριση. Όπω είπε και η κυρία Επίτροπο επίσης, ευτυχώ οι αγορές έχουν δώσει και ορισμένα θετικά σημάδια. Δεν πρέπει όμως να είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι, γιατί θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί με την αύξηση του τιμήματος του πετρελαίου που θα οδηγήσει σε αναπόδραστη αύξηση του κόστους παραγωγή στη Γεωργία. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρά τι πολιτικέ προθεσμίε, δεν μπορεί να αφήσει την Κομισιόν χωρί απαντήσει για τα θέματα αυτά. Περιμένουν πολιτικά μηνύματα η Γεωργία από το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν και γι' αυτό είναι απαραίτητο να συζητήσουμε σοβαρά αυτό το θέμα. Ελπίζω ότι η Κομισιόν θα δώσει κάποιε προτάσει, κάποιε λύσει και θα μας παρουσιάσει τις πληροφορίες που έχει και τα βραχυπρόθεσμα μέτρα με τα οποία προτίθεται να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Ο κύριος Νταντάν έχει το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που ακόμα μια φορά ήρθατε εδώ να μας ακούσατε. Η κρίση των τιμών το 2007 και 2008 τόνισε ε, το ευάλωτο των καταναλωτών απέναντι στην, ε, στις ασταθείς τιμές. Η κρίση γεωργική το 2009 νομίζω ότι πλήττει πολύ περισσότερο από ότι τα, προηγούμενα που ανέφερα τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Γιατί, Γιατί η τάση των γεωργικών τιμών ε, παρουσιαζόταν ως ε, διαρκής ε, και οι γεωργοί το 2008 και σε αρχές το 2009 έκαναν μεγάλα, μεγάλες επενδύσεις. Ε, επίσης είχαμε ούτως ή άλλως εισφορεύσει κάποια καθυστέρηση από τις αρχές δεκαετίας του 2000. Ε, πολλές φορές, κυρία Επίτροπε, είπατε ότι δεν θέλετε να παρέμβετε για να ρυθμίσετε τις, αγορά, τις αγορές. Αλλά τα τελευταία 20 χρόνια ξεχάσαμε ότι τα τρόφιμα καταρχάς είναι προσβρώσει και ότι τα χρειαζόμαστε. Ε, στα δύο άκρα της ε, διατροφικής αλυσίδας ε, θα πρέπει να υπάρχουν σταθερές τιμές. Το έχει ανάγκη ο καταναλωτής γιατί μην ξεχνάτε ότι έχει το, το νίκη, το δάνειο, την, τα σχολεία των, των παιδιών. Δεν μπορεί να πληρώνει πολλά λεφτά και για τα τρόφιμα. Επίσης, ο Γεωργός πρέπει να κάνει σημαντικές επενδύσεις αν λάβουμε υπόψη μας όλα τα τμήματα της αλυσίδας, τη μεταποίηση, τη σύντηση, ε, όλοι αυτοί μπορούν να έχουν ιδιωτικά εργαλεία σταθεροποίησης των τιμών. Κυρία Επίτροπε, μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχει διέξοδος για το μέλλον, ε, μπορείτε να συμμετάσχετε σε ένα προβληματισμό ε, γύρω από, μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ο κύριος ε, κυρία έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που ήρθατε να μας ακούσετε ακόμα μια φορά. Θα ήθελα να τονίσω διάφορα θέματα, τα οποία ήταν σημαντικά στη Βόρεια Ιρλανδία, στο γεωργικό τομέα τα, τους τελευταίους μήνες. Ίσως να διαβάσετε, κύριε Επίτροπε, ότι στην περιοχή μου είχαμε σοβαρότατες πλημμύρες ε, τις ε, τελευταίες εβδομάδες. Αυτό οδήγησε σε σοβαρότατες δυσκολίες για τους γεωργούς. Δεν μπορούσαν να αποθηκεύσουν ε, γιατί είχαν κλείσει οι δρόμοι και επιπλέον δυσκολεύονταν και λόγω της βροχής. Επίσης, δυσκολεύονται να βάλουν λιπάσματα στα χωράφια τους. Ενθαρρύνουμε την Κομισιόν να δει αυτό το θέμα και να μας πει αν μπορεί να υπάρξει άμεση βοήθεια για τους γεωργικούς μας. Επίσης θα θέλαμε η Κομισιόν να κοιτάξει τον κλάδο της πατάτας στη Βόρεια Ιρλανδία. Διάφοροι εκμεταλλευτές και γεωργοί πατάτας μου έγραψαν σήμερα γιατί επλήγησαν πολύ έντονα από τα υψηλά επίπεδα βροχοπτώσεων των τελευταίων εβδομάδων. Εκφράζουν σοβαρότατες ανησυχίες και θεωρούν ότι ε, λόγω της, του παγετού ε, και λόγω του κρύου φοβούνται ότι θα χάσουν τη σοδιά τους. Είναι ένα τμήμα της, του γεωργικού τομέα στην Ιρλανδία που αντιμετωπίζει πραγματικά μεγάλες δυσκολίες. Επίσης πρόσφατα συναντήθηκα με παραγωγούς ε, αυγών. Ε, αλλάζουν τα μεγέθη των κλοβών τους σε αυτή τη φάση και θέλουν μια εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν θα χρειαστεί να ξανααλλάξουν τους κλοβούς αργότερα. Ε, θέλουν τουλάχιστον να έχουν μια περίοδο ασφαλείας όπου αυτοί οι κλοβοί με αυτές τις διαστάσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούνται. αγαπητοί συνάδελφοι, ερχόμαστε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Έχουν ζητήσει το λόγο 7 συνάδελφοι. Σας παρακαλώ πολύ κρατήστε το χρόνο του ενός λεπτού για να μπορέσετε να παρέμβετε και οι 7. Σας παρακαλώ πολύ. Πρώτος ο κύριος Σιλβέστρης. Κυρία Επίτροπε, η κρίση του γεωργικού τομέα είναι πάρα πολύ σημαντική και μπορεί να είναι μία αναστρέψιμη. Στην απουλία ε, η γεωργία είναι η βασική οικονομική δραστηριότητα και τα εισοδήματά μας προέρχονται ε, από εκεί. Ε, έπεσε πάρα πολύ η τιμή του ελαιολάδου όμως, κατά 30 cents το εκατόλιτρο. Το παρθένο ελαιόλαδο ήταν πάντα η περηφάνεια της περιοχής μου. Αλλά νομίζω ότι έχουμε τεράστια προβλήματα. Γίνονται συνέχεια διαδηλώσεις και μπλοκ και οδοφράγματα από τους γεωργούς για τα προβλήματά τους. Ε, σας τα λέω αυτά γιατί τα γνωρίζω, τα βλέπω κάθε μέρα. Θα ήθελα να δημιουργηθεί ένα ταμείο ε, αλληλεγγύης όπως έγινε και για το γάλα. Θα ήθελα, ε, θα ήθελα επίσης αυτό να, να ισχύσει και για τα οποροκυπευτικά. Επίσης θα ήθελα να το τροποποιηθεί ο κανονισμός 2568 για τα χαρακτηριστικά των ελαίων. Επίσης θα ήθελα να να δούμε με ποιον τρόπο θα ξεσκεπάσουμε τις απάτες στα σούπερ μάρκετ ε, για να μην χρησιμοποιούν ε, λάδια διαφορετικά από αυτά που λένε ότι χρησιμοποιούν. Η κυρία Κόστιγκερ τώρα το λόγο παρακαλώ. Για ένα λεπτό μόνο κυρία Κόστιγκερ. Κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Σημαντικό το μήνυμα για τους αγρότες που προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα προστοζήν και για τις, ε, ε, ιδίως για τις προσπάθειες διάθεση των προϊόντων στην αγορά. Σε οποιοδήποτε κλάδο της παραγωγής πρέπει να διαγνώσονται έγκαιρα οι επαπειλούμενες κρίσεις και να λαμβάνονται μέτρα, ιδίως για την παραγωγή των τροφίμων. Εκεί χρειάζεται μηχανισμοί αγοράς οι οποίοι θα επιτρέψουν την διατήρηση των γεωργών στην Ήπεθρο και αυτό είναι αντικατάστατο. Όλα αυτά πρέπει να διατηρηθούν και να λαμβάνονται υπόψη στις μελλοντικέ συζητήσεις για τη νέα αγροτική πολιτική. Ο κύριος Ταραμπέλα έχει το λόγο. Σε ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τις εξηγήσεις σας ότι αφορά το κόστος διαφορών γεωργικών παραγωγών. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ε, επαγρυπνούμε, όπως είπατε, και να δράσουμε αν χρειαστεί. Ε, μιλήσατε για την αστάθεια που είναι ο, ο εχθρός νούμερο ένα της μοντέρνας γεωργίας. Θα ήθελα λοιπόν να σας κάνω έκκληση να έχουμε μια δημόσια πολιτική καθορισμού των τιμών και ρύθμισης των τιμών και στο μέλλον θα πρέπει γενικά να υπάρχει αυτή η δημόσια πολιτική ρύθμιση μέσω ενό παρατηρητηρίου ε, για τι τιμέ και τα κέρδη που θα καθόριζε ε, τι κέρδος θα έχει ο παραγωγός, ο μεταποιητής ή ο διανομέας σήμερα. Τα αφήνουμε αυτά στην, στους ιδιώτες. Συχνά όμω, ο μόνο που χάνει από όλη αυτή την ιστορία είναι ο παραγωγό. Οι άλλοι, μεταποιητή και διανομέα, κερδίζουν. Ε, και για την τιμή του, ε, ε του Η τιμή του καθορίζεται στο Σικάγο. Όμω ε, το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Όχι μόνο. Θα πρέπει να συνεισφέρουμε κι εμεί. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. <clears throat> κυρία Επίτροπε, ανησυχώ. Ανησυχώ γιατί πολλέ φορέ δεν υπάρχει συντονισμό και δεν λαμβάνει την υπόψη το κριτήριο τη αηφορίας στη Γεωργία. Δύο ερωτήματα. Πρώτον, γιατί για τη διαδικασία πιστοποίησης στη Νότια Ευρώπη με τις κλιματικές αλλαγές που είναι τεράστιες, γνωρίζοντα ότι είναι σημαντική η χρήση των εδαφών, γιατί μας δίνεται χρήματα για να ξεριζώσουμε ελαιόδεντρα, ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ερήμους εκεί που ήταν φυτεμένα δέντρα. Δεύτερον, με το Μαρόκο. Αν η Ευρώπη έχει μια εξωτερική κοινή πολιτική, πρέπει να σεβαστεί και τα συμφέροντα των πολιτών μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή γονατίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση εναντί του Μαρόκου, δεν υπάρχει καμία αμοιβαιότητα και δεν υπάρχει κανένα έλεγχο υγεία και σε ό,τι αφορά τη χρήση παρασυτοκτώνων στις χώρες αυτές παραγωγή όπω το Μαρόκο. Ανοίγοντα λοιπόν την πόρτα σε προϊόντα πέραν Τη ποσόστοση δημιουργείται και προβλήματα ποιότητα. Τώρα το λόγο θα πάρει ο κύριο Γκλάτφελντερ. Σας παρακαλώ για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ. Ήταν πολύ σημαντικό να μιλήσαμε για κρίση στους διαφόρους κλάδους παραγωγής. Διότι έχουν γίνει πολλά σχέδια για το πώς θα διαμορφωθεί η στήριξη της Γεωργίας το 2013 και μετά. Αλλά ας σκεφτούμε πόσο σημαντικές και βαριές ήταν οι συνέπειες της φιλελευθερωποίησης τα τελευταία χρόνια. Ας μην κάνουμε τα ίδια σφάλματα, γιατί το κόστος της αγροτικής παραγωγής στο μέλλον θα αυξηθεί, αλλά θα χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο τη γεωργία για να σας διατροφή των αυξανόμενων πληθυσμών. Αντί να απλουστεύονται τα πράγματα για τους ε, αγρότες, γίνονται πιο περίπλοκα. Νέα μέτρα για την προστασία των ζώων, για παράδειγμα, τα οποία αυξάνουν το κόστος και βεβαίως οι ανταγωνιστές μας τρίτων χωρών δεν έχουν τέτοια μέτρα Ε, Ο πρόεδρος Μπαρόσο στα πλαίσια της ανταλλαγής απόψεων για τις κατευθυντήρες γραμμές του είπε ότι η βιωσιμότητα και η διατήρηση των ειδών είναι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τρέχουσα περίοδο. Ο στόχος αυτός λοιπόν πρέπει να περιληφθεί σε όλους τους τομείς και κράτους παραγωγής, ιδιαίτερα στην γεωργία. Επιθυμώ σήμερα εδώ να απευθύνω εμφατικά έκκληση να προωθήσετε τα μέτρα εκείνα τα οποία θα οδηγήσουν σε αυτήν την διατήρηση των ειδών και στην βιωσιμότητα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σκέλη για ένα λεπτό. Uh, Mr. President. Um, I welcome this debate. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ βλέπω πάρα πολλά αυτά τα προβλήματα να συζητούνται που δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για αυτά. Ενώ υπάρχουν και άλλα για τα οποία μπορούμε να έχουμε μία αντιμετώπιση. Ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι το θέμα της υπερβολικής ρύθμισης. Το λένε και οι γεωργοί. Αναφέρθηκε το θέμα των ε, γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. Ένα ακόμα το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η εξαγωγή ζών των ζώων. Υπάρχει κίνδυνος η ρύθμιση στον τομέα αυτό να είναι απαγορευτική για τους γεωργούς και αυτούς που εξάγουν ζώντα βοήδη. Πιστεύω μερικές φορές ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε την, ε, τις μεταφορές των ζώων που εξάγονται με τις μετακινήσεις των Ευρωβουλευτών ως προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι οι Ευρωβουλευτές οι οποίοι ταξιδεύουν περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποια, κάποια ρύθμιση η οποία δεν θα μας διώξει από τις αγορές. Όλοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν άλλες ε, <laughs> άλλε γλώσσε. Θέλω να σα ευχαριστήσω γιατί είπατε στην αρχή mercy. Ελπίζω ότι δεν ζητούσατε έλεο. Απλώ προσπαθούσατε να μου πείτε ευχαριστώ. Όχι στα ελληνικά. Στα ελληνικά είναι ευχαριστώ, εν πάση περιπτώσει. Okay. Uh, Mr. Uh, Adrover for one minute. για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε όχι μόνο είναι ανησυχητική κατάσταση στη Γεωργία, αλλά θα έλεγα ότι είναι αφόρητη. Όλο και μεγαλύτερες διαφορές υπάρχουν μεταξύ της τιμής στον παραγωγό και της τιμής στον καταναλωτή. Σε παγκοσμίο επίπεδο είναι πια μια ουτοπία να μιλάμε για συμφωνίες οι οποίες δεν τηρούνται πλέον. Με την κατάσταση στο τομάτας από το Μαρόκο βλέπουμε καταστάσεις που ίδια η υπηρεσία κατά του, των ατασταλιών και των απατών της δακτυλοδεικτή οι κανόνες οι φυτιογειονομικοί εφαρμόζονται μεροληπτικά πολλές φορές. Υπάρχει μείωση των δασμών για τις μπανάνες που θα οδηγήσει σε πάρα πολύ αρνητικέ συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονός ότι οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το κόστος των ζωοτροφών. Όλα αυτά λοιπόν θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο την γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδίω στι υπερπεριφερειακέ περιοχέ τη Ευρώπη δεν υπάρχει μοναχά βεβαιότητα, αλλά πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Οι γεωργοί θέλουν να συνεχίσουν αυτή τη δραστηριότητα. Κάθε μέρα είναι όλο και πιο δύσκολο. Η Κομισιόν θα πρέπει να κατανοήσει τη σημασία αυτού του τομέα χωρί κανένα σύμπλεγμα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ντόρφμαν για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμες Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. όντω κρίση σημειώνεται σε πολλού κλάδου τη παραγωγή τη γεωργική πολιτική και αυτό οφείλεται εν μέρη και στα μέτρα φιλελευθερωποίηση των τελευταίων ετών. Εφόσον αφαιρούμε όλο και περισσότερα δίχτυα ασφαλείας από την αγροτική παραγωγή, τόσο περισσότερο θα διακυμαίνονται οι τιμές και θα προκαλούν προβλήματα στους παραγωγούς. Πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποιες λύσεις στα πλαίσια τη αναδιάρθρωση τη γεωργική πολιτική πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ανακόψουμε αυτέ τι διακυμάνσει των τιμών. Μετά από την θέση σε ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα, εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε το καθήκον να δραστηριοποιηθούμε. Ακόμα και αν τι τελευταίε μέρε συναντήθηκαν στο Παρίσι οι Υπουργοί Γεωργία εκτό ε, Συμβουλίου, αυτό βεβαίω είναι θετικό βήμα. Αλλά νομίζω, κυρία Πρόεδρε και κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε το καθήκον εμεί εδώ ω Ευρωβουλευτέ να δείξουμε και ποιον ρόλο θα παίξουμε, ποιον νέο ρόλο θα παίξουμε εμείς εδώ, να το δείξουμε αυτό στους αγρότες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, και τώρα για τη λήξη συζήτηση, τον λόγο έχει ε, εξ ονόματος της Επιτροπής η κυρία Φίσερ Μπόρν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις που σας που άκουσα. Η συζήτηση αυτή πάντως δείχνει σαφώς ότι υπάρχει συμφωνία ότι ο γεωργικός τομέας αντιμετωπίζει τρομερές δυσκολίες. Καταρχάς, με εξέπληξε το γεγονός ότι άκουσα ότι δεν θα έπρεπε να... ότι μάλλον αφαιρέσαμε το δίκτυο ασφαλείας. Δεν, δεν είναι σωστό αυτό. Υπάρχει το δίκτυο ασφαλείας. Σε περιπτώσεις όπου οι γεωργοί χρειάζονται υποστήριξη, το έχουμε με τις άμεσες πληρωμές. Υπάρχει λοιπόν Και επίσης έχουμε τα διάφορα συστήματα παρέμβασης, ε, ιδιωτική αποθεματοποίηση, σύστημα εξαγωγικών επιστροφών. Λειτουργούν αυτά τα συστήματα και καταφεύγουμε σε αυτά όταν χρειάζεται για την απλούστευση, για την γραφειοκρατία. Συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να εξομαλύνουμε την κατάσταση για τους γεωργούς όσο μπορούμε. Και γι' αυτό ακριβώς την Τετάρτη στη συνάντηση του Συμβουλίου θα παρουσιάσω στη Σύνοδο των Υπουργών κάποιες προτάσεις απελευθέρωσης τις οποίες θα συζητήσουμε. Το Συμβούλιο παρουσίασε 39 διαφορετικέ προτάσεις και εμείς μπορούμε να δεχτούμε κάποιες από αυτέ. Κάποιες είναι πιο πολιτικές και αφορούν την περίοδο μετά το 2013. Αλλά είμαι σίγουρη ότι τις προτάσεις αυτές θα τις ε, διαβάσετε και θα δείτε ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Όσοι μίλησαν για το θέμα των φόμικρων, συμφωνούμε απόλυτα για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, θέλω να σα πω. Είναι πολύ σημαντικό να βρούμε μια λύση για την ε, ύπαρξη μη εγκεκριμένων γάμματα φόμικρων. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε επί ενός αριθμητικού στοιχείου. Τι ποσοστό μπορεί να περιέχεται. Είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος ε, εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων. Ταυτόχρονα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και μεγάλος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε ε, πολύ καλά εμπορικά πολύ καλά προϊόντα, θεωρούνται τα προϊόντα μας πολύ ποιοτικά στο εξωτερικό και στις ε, αγορές στο εξωτερικό. Νομίζω ότι η ιδέα του να προστατεύσουμε τη δική μας παραγωγή θα ήταν καταστροφική για τη Γεωργία. Θα πρέπει αντίθετα να ανοιχτούμε στις εξωτερικές αγορές, να είμαστε ορατές, ορατοί προς αυτές και ελπίζω ότι στο μέλλον θα υπάρξει πλήρης υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για την προώθηση των προϊόντων υψηλής ποιότητας στις ε, νέες και στις αναδυόμενες αγορές. Μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερα, αν έχουμε την υποστήριξή σας. Για το θέμα του κανονιστικού πλαισίου. Δεν άκουσα ακριβώς αυτή τη φρασιολογία, αλλά νομίζω ότι αυτό εννοούσατε με τα διάφορα σχόλιά σας. Σήμερα μπορούν οι γεωργοί να συνάψουν συμβάσεις με τη βιομηχανία ειδικά στα γαλακτοκομικά, για κάποιο συγκεκριμένο όγκο προϊόντων με σταθερή τιμή. Αυτό υπάρχει ως δυνατότητα για τους γεωργούς. Και στην ομάδα υψηλού επίπεδου για τα γαλακτοκομικά εξετάζουμε διάφορους εθελοντικούς τρόπους για να βελτιώσουμε αυτό το σύστημα. Βιοπικιλότητα. Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα και ακριβώς γι' αυτό συμπεριλάβουμε τη βιοποικιλότητα στις νέες προκλήσεις όταν ε, συμφωνήσαμε για το διαγνωστικό έλεγχο τη γεωργική πολιτική τον Νοέμβριο του 2008. Αυτό λοιπόν είναι υψή τη προτεραιότητα και συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλια που ακούστηκαν από το συγκεκριμένο βουλευτή που μίλησε γι' αυτό. Για τα μέτρα τώρα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά νέες πρωτοβουλίες δεν μπορούν να παρουσιαστούν από μια υπηρεσιακή εντό αγωγικών ε, επιτροπή. Φυσικά θα το ξέρετε αυτό. Ξέρετε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, υπάρχει αυτό το κόλλημα. Επομένω, ελπίζω ότι με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν αρχίσει να λειτουργεί, θα ανοίξουν όλε αυτέ τι δυνατότητε. Γι' αυτό θέλω να ξεκινήσει να λειτουργεί το, συντομότερο δυνατόν. Με μεγάλη χαρά επίσης βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι σημαντικός παίχτης, σημαντικός εταίρος στο μέλλον. Με την διαδικασία της συναπόφασης χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν πρόκειται μόνο για συναπόφαση για τα καθαρά γεωργικά θέματα, αλλά και για τα δημοσιονομικά της γεωργίας. Θα έχετε τεράστια επίδραση εδώ. Μπορείτε να επηρεάσετε τις δημοσιονομικές δυνατότητες της γεωργίας για την περίοδο μετά το 2013. Και ίσως εγώ ε, μπορεί να μην το δω από αυτή τη θέση του Επιτρόπου Γεωργίας, θα έχω τα μάτια μου στραμμένα πάνω σας όταν αναλάβετε τις νέες σας αρμοδιότητες για τη Γεωργία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Η συζήτηση έληξε. Προχωράμε τώρα στην προφορική ερώτηση προοπτικές αναπτυξιακής ατζέντα της Δόχα μετά την 7η Υπουργική Διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Το λόγο έχει για πέντε λεπτά ο συντάκτης ερώτησης ο κύριος Μορέιρα.